παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντίας Ντεμέρα. Ευχαριστώ. Θέλω να προσπίσω τα συμφέροντα 85 εργαζομένων της επιχείρησης Ινδούστριας Λάκτεας Βάγης Ολετάνας. Είναι μια επιχείρηση με κύκλο αισιών πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ κέρδος το 2014 και πάνω από 94 εκατομμύρια λίτρα παραγωγή το χρόνο. Ε, μαζικές απολύσεις για οργανωτικούς λόγους, αλλά όχι για οικονομικούς λόγους, διότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα. Πρόκειται για μια επιχείρηση ε, μετεγκατάστασης ε, της, ε, του εργοστασίου για να μειωθούν τα κόστη. Για ποιο λόγο. Γιατί η επιχείρηση αυτή ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα κέρδη παρά για τους εργαζόμενους. Ε, ούτε καν διάλογο δεν κάνουμε τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λόγο ζητώ από την Κομισιόν να λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου να αποφύγουμε τέτοιου πρακτικές που καταστρέφουν τον επιχειρηματικό μας ιστό. Ζητώ προστασία για τους εργαζόμενους και διαφήμιση, ε, κοινοποίηση των γεγονότων. Δεν κλείνει η επιχείρηση, λένε οι εργαζόμενοι. Έτσι λέω και εγώ, δεν θα κλείσει. Τον Πιτσούλα. Ευχαριστούμε ο κύριος Πιτσούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα πάλι είχαμε μια θερμή συζήτηση για το θέμα της TTIP. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν τη φωνή τους και μάλιστα η χειρά με τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε πλέον ιδιαίτερη ευθύνη διότι εμείς τελικά λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Όμως για άλλη μια φορά ο λαϊκισμός κατάφερε αυτό που ήθελε. Ενώ ε, δυσκολεύει τι διαπραγματεύσει και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική μα θέση, διαδίδει και ψευδεί φήμε. Πρέπει λοιπόν η προστασία των πολιτών να είναι στο κέντρο των διαπραγματεύσεών μα. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά πρότυπα και η προστασία των εργασιακών πρέπει να είναι προτεραιότητα. Το ίδιο και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η προστασία των ε, σημάτων γεωγραφική ένδειξη, το τι θα γίνει με τα, γεωγραφικά. με γενικώ τροποποιημένα και οι διευκολύνσει θεωρήσεων για επικόστη των χωρών. Εδώ πρέπει να δείξουμε την επικοδομητική μα στήριξη στι ανάγκε των πολιτών και. Ε, με συγχωρείτε. Bilbao. Κυρία Μπιλμπάου Βαραντίκα, η Ισπανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα γιόρτασε την, Ευρωπαϊ... την Παγκόσμια ημέρα ε, ε τύπου και μέσω μαζικής ενημέρωσης με το, την πάυση με αναμετάδοσης ε, του τηλεοπτικού σταθμού της Ναβάρας μέσω του κρατικού, ε, της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Ε, το μέτρο αυτό αφορά μόνο την Αβάρα. Συνεπώ, αποτελεί διάκριση και τεχνικά είναι αδύνατο να γίνει και πολιτικά είναι ακατανόητο. Διότι οι πολίτε στην Αβάρα ε, έχουν υποστηρίξει αυτέ τι εκπομπέ. Ενώ η τεχνολογία ανοίγει ορίζοντες στην ε, πολυπολιτισμικότητα και, στην, ε, ε, στο, και στη διαφορετικότητα, γλωσσική και άλλη, κάποιοι την περικόπτουν. Ευχαριστώ. Γόνος. Ευχαριστούμε κύριος Χρυσόγονο. Τις τελευταίες ημέρες η τουρκική προκλητικότητα απέναντι στην Ελλάδα έχει υπερβεί κάθε προηγούμενο. Με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας κατοικημένων νησιών στο αιγαίο ή ακόμη και στο λιβικό πέλαγος με υπερπτήσεις σε χαμηλό ύψος πάνω από ελληνικά νησιά και με παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων. η συμπεριφορά αυτή της τουρκίας εγκυμονεί διαρκώς κινδύνους για νέα αεροπορικά ή ναυτικά δυστυχήματα <clears throat> κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων με βάση το διεθνές δίκαιο αναχαιτήσεων από τις ελληνικές αεροναυτικές δυνάμεις όπως έχει συμβεί επανειλημμένα και στο παρελθόν. το κυριότερο όμως είναι ότι η ελλάδα υποχρεώνεται έτσι σε υψηλές αμυντικές δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά της προβλήματα και αποτελούν ιστορικά μια από τις κυριότερες αιτίες υπερχρέωσης της χώρας. εφόσον η ευρωπαϊκή ένωση απαιτεί τη μείωση των ελληνικών αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του ελληνικού προγράμματος οφείλει να αναλάβει έναν αντίστοιχα πιο ενεργό ρόλο στην αναχέτηση της τουρκικής επιθετικότητας. Πέρσι προειδοποίησα για τους κινδύνους σε βάρος των παιδιών μετά τις κρίσεις. Χιλιάδες παιδιά εξαφανίζονται από διακινητές Τώρα έχουν πολλαπλαστεί οι αριθμοί και η Ιντερπολ προειδοποίησε ε, ότι εξαφανίστηκαν 10.000 παιδιά στις αρχές του χρόνου. Ε, μόνο στην Ιταλία ε, περίπου πάνω από 1.000 στη Σουηδία. Δεν γνωρίζει κανείς που βρίσκονται, τι κάνουν, με ποιον είναι. Η Άγγελα Μέρκελ και άλλοι υπέρ των ανοιχτών συνόρων είπαν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ε, αυτή είναι μία θεδιών ε, στην, στην ε, ευρωπαϊκή ιδεολογία και το Κοινοβούλιο αυτό δεν κάνει τίποτε. Ευχαριστούμε, η κυρία Τερικάμπας. Ο κύριος Τερικάμπας. Θα ήθελα με την ευκαιρία της ημέρας Ευρώπης να πω δύο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει να ε, μην είμαστε ευρωσκεπτικιστές, να είμαστε ευρωκριτικοί. Τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν μόνο με περισσότερη Ευρώπη, όχι με λιγότερη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας μεγάλο όραμα και θα πρέπει μέσω πρόθεσμα να γίνει σημείο αναφοράς για όλους. Και σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ευημερία και σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως Καταλανός θα ήθελα επίσης να πω ότι οι συμπολίτε μου είναι προσιλωμένοι στην, στο να εργαστούν στο μέλλον με την Ευρώπη στενά. Με μια Ευρώπη που θα προασπίζεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και η, Καταλούνια, η Καταλωνία μόλις πολύ σύντομα γίνει νέο ευρωπαϊκό κράτος θα συνεχίσει την συνεργασία της με την Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. 160.000 εκτάρια δάσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα μου η Γαλλία είναι η τρίτη στην επιφάνεια αυτή ε, αναλογικά. Όμω ο τομέας της ξυλίας έχει χάσει πάνω από 60.000 θέσει εργασία τα τελευταία 10 χρόνια και τα υλοτομία ή ε, τα, οι μονάδε επεξεργασία ξύλου ε, κλείνουν. Η, στη, στο Μοζέλα έχει κλείσει εργοστάσιο πρόσφατα με 3.000 θέσει εργασία να χάνονται. Αυτά τα θλιβερά αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα του ντάμπινγκ τη Κίνα προ την οποία ε, με εξευτελιστικέ τιμέ εξάγουμε τα πρώτα ξυλία μα ε, πρώτη ύλη για να τα πάρουμε πίσω επεξεργασμένα. Τα, οι πρώτες αυτές ύλες, όπως ε, τα ξύλα που παράγονται στην Ευρώπη, θα έπρεπε να, να είναι αντικείμενο επεξεργασία κοντά στον τόπο παραγωγής τους, όχι στην ελέγχη του πλανήτη για να ξανάρχονται ως έτοιμα τελικά προϊόντα. Είναι πολλοί αυτοί που εξάγουν τα προϊόντα τους προς την Κίνα αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει αυτές τις πρακτικές ε, λόγω αυτού του υπερφιλελεύθερου dumping. Θα πρέπει να δούμε ότι πλήττονται οι θέσεις εργασίας σε εμάς και ότι ο πλανήτης αποδυναμώνεται. Ευχαριστούμε πολύ ο κ. Ζαριανόπουλος. Αποφασίσετε σαν Ευρωκοινοβούλιο να μετονομάσετε τη σημερινή επέτειο την 9η του Μάη από μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών σε μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γέννημα των μονοπωλίων ξαναγράφετε την ιστορία εξισώνοντας τον φασισμό με τον κομμουνισμό κλιμακώνοντας τον αντικομμουνισμό στηρίζοντας τις διώξεις κομμουνιστών σε πολλές χώρες στείνοντας φιέστες και σπίτια παραχάραξης της ευρωπαϊκής ιστορίας. αντικειμενικά καλλιεργείται έδαφος για την αναβίωση του φασισμού που γεννά σαν εφεδρεία η καπιταλιστική σύψη και βαρβαρότητα. ούτε την ιστορία μπορείτε να αλλάξετε ούτε τη λαϊκή μνήμη να σβήσετε τιμάμε όσους πολέμησαν με κάθε τρόπο τον ναζισμό φασισμό τότε και τώρα. τα κομμουνιστικά κόμματα που ηρωικά ηγήθηκαν των εθνικοαπελευθερωτικών και αντιφασιστικών κινημάτων τον τιτάνιο αγώνα και θυσίες της σοβιετικής ένωσης εκατομμυρίων μπολσεβίκων και σοβιετικών ανθρώπων που κάρφωσαν την κόκκινη σημαία στην καρδιά του ναζιστικού θηρίου στο Ράιχσταγκ. η ιστορία δεν πισωγυρίζει. ο 21ος αιώνας είναι η εποχή νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων για την κοινωνική απελευθέρωση.

Σήμερα γιορτάζουμε τη μέρα της Ευρώπης και κάθε χρόνος με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να είμαστε περήφανοι για αυτά που πετύχαμε και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Φέτος όμως έχουμε πολύ άριθμα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε που δεν φαίνεται να έχουν κατάλληλες λύσεις και δεν υπάρχει και καμία αλληλεγγύη. Ο καθένας από εμά στην Ευρώπη πρέπει να δει τι χρειάζεται να αλλάξει προκειμένου η Ευρώπη να επιβιώσει. Συζητάμε σημαντικά θέματα όπως ε, η μετανάστευση, η οικονομική κρίση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα ε, πράγματα που θα πρέπει να μας απασχολούν και άλλα πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό. Τα συμπληματικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Νομισματικής Ένωσης δεν εξαρκούν. Πρέπει να προσέξουμε κάθε κατός μέλος να τηρεί τους κανόνες αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη. Πρέπει να προχωρήσουμε να γίνουν οι διαφθορτικές που τόσο χρειαζόμαστε. Είναι τόσο δύσκολο αυτό, αλλά αν το κάνουμε θα έχουμε νομίζω πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Ε, Ντάντζελα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρω... απελευθέρωση του καθεστώτο ε, των θεωρήσεων για του πολίτε τη Γεωργία που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ώρα που ε, απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση τη προόδου τη Γεωργία και του κράτου τη, τη ε, μεταρρυθμίσει που πρέπει να υλοποιήσει για να προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι ότι όσα έχουν εξαγγείλει στη Γεωργία είναι πράγματα που τώρα στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω το το κοινοβούλιο και τα κάτι μέλη πρέπει να στηρίξουν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί όντω υπάρχουν βήματα πρόοδου στη Γεωργία. Και η Αρμενία στηρίζει. Η Ρουμανία μάλλον στηρίζει τις ε, φιλοδοξίες της Γεωργίας ε, στην ε, προσέγγισή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν σημειώσει τις θετικές εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση της ε, Γεωργίας και θα πρέπει να επιτύχει πλήρως και τα κριτήρια που ορίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες ε, του λαού της Γεωργίας για το θέμα αυτό και καλό θα είναι κάποια στιγμή να δώσουμε μια ενθάρρυνση. Ευχαριστούμε, Ράντος Γιώργο. Ευχαριστώ. Οι ορεινές ε, απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ενεργειακή ένδια και κρίση. Ένα σύμπτωμα είναι η χαμηλή ενεργειακή απόδοση στα κτίρια γραφείων και στα διαμερίσματα. Ε, είναι δεδομένων των αυξημένων δαπανών ε, επιδεινώνεται η κατάσταση. Θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αναπτύξει προγράμματα μέσα στα υπάρχοντα, στα υφιστάμενα ταμεία για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ώστε οι διαδικασίες ε, για τη χορήγηση κονδυλίων να πλουστευτούν και να γίνει και μια ενημερωτική εκστρατεία ώστε οι ντόπιοι συντελεστές να ενημερώνονται καλύτερα και να χρησιμοποιούν την διαθέσιμη χρηματοδότηση καλύτερα. Έτσι, η ενεργειακή απόδοση θα μπορέσει να αναβαθμιστεί και θα βελτιωθεί και το επίπεδο ζωής τους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λόπες. Κυρία Λόπες Βερμέχο. Ε, γιορτάζουμε 71 χρόνια από τη νίκη εναντίον του φασισμού στην Ευρώπη 71 χρόνια από τη νίκη των ε, λαών και της δικαιοσύνης η Ισπανία αποτέλεσε θύμα του ψυχρού πολέμου με το Φράνκο και έγινε πιόν της ιστορίας. Όμως χαιρέτησε αυτή την νίκη με την ίδια χαρά και αγαλίαση. Με τον ίδιο πόθο να ζήσει σε δημοκρατία και δικαιοσύνη. Όμως σήμερα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη προδίδει την ερωτική της τάξη που τους αρνείται την αξιοπρέπεια και το ψωμί, που αρνείται την είσοδο στους μετανάστες και δίνει τροφή στα τέρατα τα οποία υποτίθεται ότι καταπολεμάει. Δίνει λαβή για την ανάπτυξη μιας ακροδεξιάς. Θα ήθελα να διεκδικήσω τη μνήμη αυτών που εργάστηκαν κατά, ε, πολέμησαν κατά του φασισμού. Οι αγώνες τους ε, είναι παρόντες περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ε, στο δρόμο, στα σπίτια, στις στην εργασία θα πρέπει όλοι μαζί η εργατική τάξη να σηκώσει το ανάστημά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μόη. Δεν είναι. Ο κύριος Λεμπρετών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Επίτροπος Μοσχοβεσί επιβεβαίωσε ότι οι πρόσφυγες στηρίζουν την ανάπτυξη. Κατά την άποψη της υποδοχή των προσφύγων θέλει είναι ένας λόγος και ένα κίνητρο οικονομικής ανάπτυξης θα φτάσει το 2% στην Ευρωζώνη το 2016. Εκτιμά ότι οι δημόσιες δαπάνες υπέρ των προσφύγων παράγουν ένα 0,30% ε, ε, του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 0,25% συγκεκριμένα στη Γερμανία ως προς το ΑΕΠ και την ανάκαμψη. Οι μελέτε όμω και τα πορίσματά του τα τελευταία χρόνια δείχνουν τι καταστροφικέ συνέπειε τη μετανάστευση για την Γαλλία συγκεκριμένα. Μια μελέτη του 2012 του Ζαν Μπολ Κούρεβιτ δείχνει ότι το κόστο στον προπολογισμό είναι 17 δι του ευρώ και του κυρίου Μποζακόφ το 17, 84 δι ευρώ ε, πλέον, επιπλέον κόστος λόγω των προσφύγων, είναι δικαιοσύνη, το κοινωνικό σύστημα, την υγεία και την πρόνοια, τη στέγαση. Το συμπέρασμα είναι ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Βρυξελών ψεύδεται ασύστολα ενώπιον των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρόλα. 23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. 76 εκατομμύρια εκατομμύρια δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Ανθρώπινο δράμα. Το κοινωνικό μας ε, σύστημα ε, παραπατάει. Το, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ε, υποστηρίζει ένα καινούριο πλαίσιο κατάρτισης ε, ε, που θα στηρίζει την κατάρτιση και την απασχολησιμότητα ταυτόχρονα. Ε, η μάθηση θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες που περιμένει η αγορά εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι δημόσιες αρχές και τα κέντρα κατάρτισης θα πρέπει να συνεργαστούν. Ε, το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ε, επιτρέπουν να προχωρήσουμε και μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την κοινωνικο-επαγγελματική επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται θετικά σχέδια και οράματα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στην Ισπανία εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και η μόνη απάντηση που βρήκε η Ισπανική κυβέρνηση ήταν η παθητικότητα, η αδιαφορία. Χιλιάδες άτομα επίσης ε, υφίστανται καταχρήσεις από όρους στα ενυπόθηκα δάνειά τους. Ε, οι δικαστές δεν μπορούν να απαγορεύσουν την ε, πώληση ενός ε, μιας οικίας οικογένειας ε, που έχει εκδιωχθεί από το σπίτι της επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειό της μέχρι ότου να εξεταστούν οι όροι της σύμβασης του ενυπόθηκου δανείου. Θα ήθελα η Κομισιόν να παρέμβει και να δώσει μια λύση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ άσχημες οι ειδήσει από την ε, παρακολούθηση της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία. Φαίνεται ότι υπήρξαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και εκδηλώσεις βίας κατά μήκος της γραμμής των συνόρων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Ε, πρόκειται για σαφείς παραδιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία με, μετά την τριμερή συνάντηση διασφαλίζει την κατάπαυση του πυρός αλλά Τώρα θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να κατησχίσει η κατάπαυση του πυρός, γιατί οι όσοι κατοικούν στην περιοχή αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και ανθρωπιστική κρίση και οι ανταποκριτές που επιστρέφουν ε, λέγουν ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ο κύριος Κάρθη. Δεν είναι στην αίθουσα. E- Ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια κρόαση για τις τραπεζικές εργασίες δημόσιες ιδιωτικές. Ε, αναφέρθηκαν διάφορες διαδικασίες για να ε, υπάρχει και ένα σύστημα παρόμοιο στην Ιρλανδία με συνεργασία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν υπερβολικό έλεγχο της οικονομίας, ιδιαίτερα με τα υψηλότατα επιτόκια που έχουν. Πώς γίνεται να υποστηρίζουμε τις τράπεζες αυτές που κλέβουν τόσα πολλά χρήματα χωρίς να δίνουν στους απλούς ανθρώπους ωφέλη. Ε, είμαστε υπέρ τη δημόσιας τραπεζικής ε, εστιάζουμε σε πραγματικές αλλαγές και στην υποστήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την κοινωνική οικονομία, του συνεταιρισμούς. Πρέπει να αρχίσει η αλλαγή και να γίνει άμεσα. Η κυρία Φων Στόρκ. Το Συμβούλιο της ε, Κεντρικής Τράπεζας στην παντοδυναμία του ε, κατάργησε το ε, νόμισμα των 500 ευρώ γιατί χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ε, ενεργειών, ξέπλυμα χρημάτων. Δηλαδή θα καταπολεμηθεί το έγκλημα αποσύροντας το, τα 500 ευρώ και αντικαθιστώντας τα με 200 συν 200 συν 100 Πώς είναι δυνατόν. Η νομισματική πολιτική είναι σημαντική. Η έκτη και ο Μάριο Ντράγκη πρέπει να ε, ε, ε, ασχοληθούν με τα αρνητικά επιτόκια. Διότι αυτός ο οποίος δεν έχει να περιμένει επιτόκια από την τράπεζα θα τα αποσύρει και θα τα κρατήσει ρευστά. Το, τα ρευστά θεωρούνται ότι είναι ελευθερία. Και όσοι θέλουν να κατακαταργήσουν, ε, θεωρούνται ε, ολοκληρωτικοί. Ο κ. Μπόκοβιτς. Πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε την ε, εναρμόνιση των θέσεών μας για την ένωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κομισιόν και των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Εμπορίου. Ατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Τις τελευταίες μέρες, πριν από μερικές μέρες, ακούσαμε ότι η, η Greenpeace ε, αποκάλυψε κάποια... Ε, ε, μάλλον υπέβαλε κάποια πληροφορίε σε ένα ανεπίσημο έγγραφο το, τις οποίες η Κομισιόν δεν κατάφερε να λάβει υπόψη. Ε, χρειάζεται διαφάνεια γιατί η αδιαφάνεια είναι ο μεγαλύτερο εχθρό αυτών των συμφωνιών. Θα ήθελα να καλέσω την Κομισιόν ε, να προσπαθήσει να ε, λάβει υπόψη τις ιδιαίτερα τις ανάγκες ε, της ασφάλειας των, ε, ασφάλειας των πολιτών και να μην βασίζεται σε κρυφά έγγραφα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Ward. Ευχαριστώ. Στις 9 Μαΐου, ακριβώς πριν από 66 χρόνια, η διακήρυξη των διευθυντών του ανθρώπου ε, ξέφραζε μια, ένα όραμα για την ειρήνη και την ανθρωπότητα στην Ευρώπη μετά από τη συντρίμια του πολέμου. Αυτά ήταν τα ιδρυτικά θεμελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 9 Μαΐου, μέρα της Ευρώπης, και πάλι βλέπουμε γενοκτομίες, εγκλήματα πολέμου και εχθροπραξίες στα σύνορά μας, με ξενοφοβία και ρατσισμό να εντείνονται σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να φανούμε συνεπείς με την ιστορική μας κληρονομιά και να εκφράσουμε σαφείς πολιτικές προτεραιότητες, να αναλάβουμε δράση για να πάψουν οι φρικαλαιότητες και οι γενοκτονίες όλο τον κόσμο το κίνημα κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη ε, πριν από κάποια χρόνια προσπάθησε να έρθει σε επαφή με βουλευτές ανά την Ευρώπη για να αναλυθεί δράση για τη Βοσνία και την Αρμενία και να διδαχθούμε από τα αποτελέσματα του παρελθόντο. Πρέπει αυτή την τραγική ιστορία να τη χρησιμοποιήσουμε ως πλατφόρμα για το διαπολιτισμικό διάλογο και τις ε, ανταλλαγές μας. Ποτέ ξανά πρέπει να πούμε.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 krajem Υπήρχαν προβλήματα τέλος Απριλίου με, τον παγετό και στην Κροατία πολλές εισοδίες κατεστράφησαν σχεδόν ολοσχερός. Ε, υπήρχαν πάρα πολλές ζημιές φρούτων, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχαν ε, καταστροφές και στην Ουγγαρία, την Αυστρία και μετά την ε, τελευταία ε, κρίση που έπληξε, του εμπάργου που έπληξε τους φρουτοπαραγωγούς, ο παγετός είναι ένα νέο πλήγμα που θα τους αποτελειώσει αν ε, βοηθήσουμε δραστικά. Ε, κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει να, αντιμετωπιστεί, να, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους οι πληγέντες από αυτό το φυσικό φαινόμενο. Η, η υποστήριξη αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχιστεί η παραγωγή οποροκυπευτικών και να προστατευτούν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Η κυρία Άντερσεν. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ε, παράδοση, την εξέλιξη των υπηρεσιών ε, των ταχυδρομείων και υπηρεσίας, υπηρεσιών δεμάτων. υπάρχουν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προστατεύουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου περί του χειρισμού ταχυδρομείου και δεμάτων. Οι κανόνες δεν απαιτούν ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομείων ε, που ε, ε, προσφέρει θέσεις εργασίας αλλά και τεχνολογία. Τα φυσικά προϊόντα χρειάζονται να φτάνουν σε εμά. Πολλά εκατομμύρια θέσεις εργασίας υπάρχουν στον τομέα των ταχυδρομείων και των υπηρεσιών θεμάτων. Εμείς θέλουμε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην γίνουν επισφαλείς. Ε, Επίση και εγώ και πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάνω από 50, ε, είμαστε υπέρ τη σχετική εκστρατεία, ούτω ώστε να αποφασίζει ο κόσμο σωστά για το πώ θα λαμβάνει βασικέ πληροφορίε που επηρεάζουν τη ζωή του. Να μα υποστηρίξετε, παρακαλώ, ε, στην εκστρατεία αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και 65 χρόνια το όραμα για την ασφάλεια στην Ευρώπη εξαγγέλθηκε από τον κύριο Σούμαν 5 χρόνια, 15 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Προσπαθούσε να συνέλθει από τις ουλές και τα τραύματα του πολέμου. Ήπειρος. Δεν θέλουμε λοιπόν να ξαναζήσουμε τις ίδιες φρικαλαιότητες. Είπε ο κύριος Σούμαν ότι τα θεσμικά όργανα μιας νέας αρχής και η Ένωση Γαλλίας και Γερμανίας μαζί με τις υπόλοιπες χώρες θα συμμετάσχουν είναι μια πρόταση που θα επιτρέψει να έχουμε την πρώτη έδρα μιας Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αναγκαίας για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Εδώ πριν από 65 χρόνια ήταν ήδη σαφές ότι ο δρόμος για την ασφάλεια της Ευρώπης δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Νομίζω ότι καλό είναι να το θυμόμαστε. Έτσι κι αλλιώς στην Τσεχοσλοβακία είχαμε όνειρα ε, τα οποία αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε να τα ζήσουμε. Οι, οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν αυτή την τόλμη στο παρελθόν για να την ξαναέχουμε κι εμείς τώρα. Ε, θα αναφερθώ στην επιστροφή περιουσιών στη Ρουμανία. Διάλεξα αυτό το θέμα διότι πρόσφατα ένας Ούγγρος Ευρωβουλευτής ε, κατηγόρησε τη Ρουμανία ότι επιβάλλει διακρίσεις εναντίον της Ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία ε, η Ρουμανία, θα ήθελα να σας πληροφορήσω, όπως και όλες οι άλλες πρώην κομμουνιστικές ε, χώρες, ε, ε, ξεκίνησε τις επιστροφές μετά το 1990. Η διαδικασία ήταν πολύ δυσχερή. Στον Ιανουάριο του 1993, 3 εκατομμύρια άτομα... Ε, ζούσαν σε εθνικοποιημένα κτίρια. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη ζωή τους. Ε, πολλοί από αυτούς ήταν γέροντες, ε, ηλικιωμένοι. Η διαδικασία ήταν δύσκολη, διότι δεν υφίσταν το πολλά έγγραφα που να πιστοποιούν το καθεστώς, το προσιακό καθεστώς πριν της εθνικοποίησης. Σε μια μικρή πόλη, στην Αγιούτ για παράδειγμα, ένα, ένα κτίριο το οποίο επιστράφει στην εκκλησία ε, έθεσε σε κίνδυνο την ε, ζωή μιας οικογένειας γιατί της κόπηκε το ελεκτικό ρεύμα. Ευχαριστώ. Ε, Ε, η νίκη κατά του φασισμού ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Αυτός, αυτή η μέρα εορτάζεται στη χώρα μου στις 8 και 9 Μαΐου. Ε, φανταστείτε ε, και τώρα στη Ρήγα και σε άλλες χώρες της Λετωνίας ε, εορτάζεται η πτώση του ναζισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γεννήθηκε η ιδέα της Ευρώπης χωρίς ε, σύνορα. Σήμερα θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και σε άλλους ε, ανθρώπους που ε, δεν έχουν την ηθαγένεια της ε, Λετωνίας και της Εσθονίας αλλά που θα πρέπει να συμμετέχουν στις ε, ευρωπαϊκές εκλογές. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Αύριο Τρίτη θα αρχίσουμε στις 9